Um, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε με την ε, τελική ψηφοφορία, την τελευταία για σήμερα, που θα κάνουμε με μεγάλη χαρά σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών ε, Θεμάτων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα τεστ του ηλεκτρονικού συστήματος. Να δοκιμάσουμε το σύστημα, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία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 We can start with compromise five. Those in... Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13. Υπέρ κατά αποχές. Να τα ελέγξουμε. Ελέγχουμε το 13. Άρχεται η ψηφοφορία. You're welcome. Vote is closed. Is adopted. Amendment 14 in favor. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τροπολογία 19. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε άρχιτη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 24. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τροποποιήθηκε άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 43 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά, 6 αποχές. Vote on the decision. Ψηφίζουμε την πρόταση να μπούμε σε διοργανική διαπραγμάτευση. Ε, άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. The vote Πέρας της ψηφοφορίας. 42 υπέρ, 11 κατά, 2 αποχές. Δεν έχουμε την ειδική πλειοψηφία, η οποία είναι απαραίτητη για να μπούμε σε διοργανικές και διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Άρα, θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια και πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά ε, της 24ης Μαΐου του 2018. δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ όλους. κυρίως τη λήξη της συνεδρίασης.